the Atlantic mackerel fishery, and an oral question to the Commission on the conservation of sea bass. So, I give the floor to the... Του Λιθρινίου. Να δώσω το λόγο στον ομιλητή. Ε, Αποσιάζει. Ο κύριος Γκάλαχερ έχει να παίξει με τη Λιβερπούλ. Ο κύριος Καντέκ... Κούκου. Ε, Κύριε Καντέκ. Να γαλλικά. Κάνε τα γαλλικά άμα μιλήσει. Σαν κανονική ολομέλεια. Um, Mr. Mato. Κύριος Μάτο. Εδώ, εδώ είμαι, κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι πολύ δεν είμαι οπαδός της ανάγνωσης κειμένων, αλλά είναι ειδικέ οι συνθήκες στη συζήτηση αυτή. Οπότε θα διαβάσω. Κύριε Πρόεδρε, εδώ έχουμε μια κοινή συζήτηση για το σκουμπρί και το λιθρίνι αλλά ο κύριος Καντέκ μίλησε για άλλα θέματα. Είναι ε, κρίμα που δεν είναι εδώ ο Επίτροπος Γιατί εδώ θα ήταν ε, μια ευκαιρία να τον συγχαρούμε για τη συμφωνία που πετύχαμε με τα κράτη του Βορειοανατολικού Ατλαντικού. Πάντω, είναι πολύ καλή ευκαιρία να μπορεί κανεί να κάνει μια τέτοια παρέμβαση μετά από μια ανάλογη συμφωνία, διότι η αλία του σκουμπριού δεν είναι κάτι το καινούριο. Έχουν υπάρξει πολλέ σχετικέ πρωτοβουλίε και το Ευρωκοινοβούλιο έχει δείξει εξαιρετική υπομονή ω προ το θέμα αυτό και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, κατά την προετοιμασία τη χθεσινή μου παρέμβαση, ε, με έθεσα πολλέ ερωτήσει στον εαυτό μου. Γιατί μέσα στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς δεν μπορέσαμε να πετύχουμε μια οριστική συμφωνία για, τα, για τις ποσοστώσεις. Εδώ με την αλία του σκουμπριού μπορεί να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα. Δεν θα έπρεπε να προβλέψουμε μονομερός, μάλλον η πρόβλεψη μονομερών ποσοστώσεων από την Ισλανδία και τις νήσους Φερόες είναι, χώρε, είναι κινήσει που πλήττουν την ισορροπία που έχουμε πετύχει με τι χώρε με τι οποίε συνεργαζόμαστε. Υπάρχουν λοιπόν κάποιε χώρε που δεν σέβονται του κανόνε. Ενώ κάποιε άλλε πρέπει να υποστούν τι συνέπειε και μάλιστα πολύ αυστηρέ. Γιατί να υπάρχουν λοιπόν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρόντουστ έχει κατόπιν το λόγο. Μόλις μπήκε βλέπω. Δεν είστε, τρέχουμε λέμε. Είστε κάτι μου λένε εδώ πέρα. Με ειδοποιούν ότι είστε. Okay, sorry. A case of mistaken identity. Α, λάθος, με συγχωρείτε. Συμβαίνουν αυτά. So, I give the floor to Mrs. Bilbao Barandica. Ο λόγος στην κυρία Bilbao Barandica. Να συγχαρώ και εγώ την Επιτροπό Δεμανάκη για αυτή την ε, νέα συμφωνία με την Νορβηγία και τις νήσους Φερόες. Όμως χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη συμμετοχή καθώς και επιστημονική ε, σχολαστικότητα για να έχουμε και μια ανάλογη συμφωνία με την Ισλανδία. Δεν μπορεί η Ισλανδία μόνο μερός να συνεχίσει να αυξάνει τις ποσοστώσεις της. Όταν ε, υπήρξαμε μάρτυρες στο γεγονότο το 2006 με τις ποσοστώσεις της Ισλανδίας να αυξάνονται για τρία είδη όπως ε, η ίδια θεώρησε σωστό, αυτό οδήγησε σε προβλήματα για τον ευρωπαϊκό στόλο και για την βιώσιμη ελεία γενικότερα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την Ισλανδία να αποφασίσει αν θα προβλέψει κυρώσεις. Η Ισπανική κυβέρνηση Η Ισπανική κυβέρνηση έχει ανάγκη και εκείνη από ποσοστώσεις, οι οποίες με αυτές τις μονομερείς κινήσεις δεν μπορούν να εξασφαλιστούν. Ευχαριστούμε, η κυρία Κούλμα. Κύριε Πρόεδρε, αν δούμε το 2009, το μικρόφωνο της ομιλήτριας όμως δεν μπορούμε να δουλέψουμε υπ' αυτές τις συνθήκες. Βεβαίως, αντικείμενο της ε, διαπραγμάτευσης ήταν τα δικαιώματα που είχε η ίδια η Ισλανδία, δηλαδή η ζώνη αποκλειστικής αλληλείας ε, του 2009. Το μικρόφωνο της ομιλήτριας ε, έχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να εργαστούμε από αυτές τις συνθήκες.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 είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε με την Νορβηγία και να ξεκαθαρίσει το τι γίνεται με το σκουμπρί, τις ποσοστώσεις ε, εκεί όπου έχουμε κοινέ αλλιευτικές ζώνες, ε, στην Σκαγεράκη και σε διάφορες άλλες ζώνες. Τώρα, αν συμφωνήσουν οι Νορβηγοί έχει ανοίξει ο δρόμος για μια νέα συμφωνία. Έτσι μπορεί να πιστοποιηθεί και η ρέγγα της ε, Βαλτικής ε, σύμφωνα με το MSE. Έτσι μπορεί να ε, πουλήσουμε αυτό το ψάρι και βεβαίως και οι ψαράδες του Μεκλεμβούργου και της Άνω Πομερανίας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Thank you very much, uh, Mr. Kuhn. The next speaker is Mr. Ευχαριστούμε, κύριος Μιλάνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε τους συντάκτες της έκθεσης. Ελπίζουμε ότι οι συνάδελφοι στη νέα ότι θα ξεκινήσει μια νέα εποχή για να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα, γιατί ο κανονισμό αυτός αφορά θέματα ουσίας. Εδώ μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα, είδαμε μια νέα ε, αρμοδιότητα για το Κοινοβούλιο, που όμω δεν εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση ε, για το Κοινοβούλιο με τη συναπόφαση, με τη διαδικασία τη συναπόφαση. Ο κανονισμό αυτό, κατά την άποψή μου, δεν είναι σωστά ε, φτιαγμένο. Θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο κανονισμό για του ελέγχου, κάτι που εύχεται και το Κοινοβούλιο και θα εξυπηρετήσει και τα κράτη-μέλη, προκειμένου να υπάρχει μια πολιτική με περισσότερο περιφερειακή διάσταση και να έχουμε μια σωστή παρέμβαση για να πετύχουμε τους στόχους μας. Είναι υπερησιόδοξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, αλήθειες αυτές συμφωνίες. Η πολιτική συμφωνία ε, είναι κάτι που τέθηκε σε κίνδυνο από τις τεχνικές λεπτομέρειες και η πολιτική διάσταση του θέματος για μας είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ε, υποβαθμίζουμε. Και για μένα λοιπόν και για την ομάδα μου αυτό συνεχίζει να αποτελεί μια προτεραιότητα. Ευχαριστούμε κύριε Μιλάνα. Ο κύριος Μπούζεκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή βεβαίως είναι η βάση ολόκληρης της ε, εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τα απαλέτητα μέσα στη διάθεσή της, ε, αλλιώς οποιαδήποτε συζήτηση δεν έχει κανένα νόημα. Μόνο μία οικονομική και οικολογική ε, αλλαγή είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε συχνά υπάρχουν και μεταναστεύσεις ψαριών και βεβαίως η προστασία των ειδών αυτών πρέπει να είναι πραγματική όχι μόνο στο επίπεδο των δηλώσεων γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω να δώσει κίνητρα στις αλληλευτικές εταιρείε ε, να χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους εκείνες που επιτρέπουν την καλύτερη επιλογή που υπάρχει σήμερα στην αγορά για να μειωθεί ο όγκος των απορρίψεων. Συνελώντη υπήν, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε... Κοιτάξτε, εγώ όσο ήμουν Ευρωβουλευτής ε, ήμουν υπέρ της ε, αλληλείας με αυτόν τον τρόπο και θα συνεχίσω. Ο κύριος Δανέλης έχει κατόπιν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Μάισνα για την εξαιρετική συνεργασία και να τη συγχαρώ για την πολύ καλή έκθεση. Η οδηγία για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών είναι ένα εργαλείο καταλητικής σημασίας για την υλοποίηση της γαλάζιας ανάπτυξης. Οι νέοι θαλάσσιοι κλάδοι που αναδεικνύονται τα τελευταία χρόνια είναι έτοιμοι να συμβάλλουν στην πολυπόθητη οικονομική μεγέθυνση, να συνεισφέρουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας και μάλιστα νέες. Οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιοτεχνολογία, οι εξελιχμένες μορφές τουρισμού είναι μόνο μερικές εξ αυτών. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η οδηγία θα απλοποιήσει και θα διευκολύνει τις επενδύσεις ειδικά αυτές που αφορούν διασυνοριακές θαλάσσιες περιοχές. Αν δεν εφαρμόσουμε ένα συνεκτικό σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού, ώστε να οριοθετηθούν σε κάθε ευρωπαϊκή περιφέρεια οι θαλάσσιες χρήσεις, η γαλάζια ανάπτυξη δεν μπορεί να υποστηριχτεί. Η άναρχη και ταυτόχρονα ανάπτυξη πολλών δραστηριοτήτων στη θάλασσα και τις ακτές απειλούν το ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον ένα περιβάλλον το οποίο τουλάχιστον στη Μεσόγειο βρίσκεται ήδη υπό τεράστιες ανθρωπογενείς πιέσεις. Γι' αυτό άλλωστε θέλουμε τους στόχους οδηγίας να διατυπωθεί ξεκάθαρα η χρήση της προσέγγισης του οικοσυστήματος αλλά και η γενικότερη πλαισίωση της θαλάσσιας χωροταξίας από μέτρα για τις παράκτιες ζώνες. Επιπλέον, από την πλευρά των σοσιαλιστών τονίσαμε την ανάγκη συνεργασίας σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης. Στην τελική της μορφή, η έκθεση ζητεί από γειτονικά κράτη να στοχεύσουν σε ένα κοινό όραμα για τον καταμερισμό των θαλάσσιων χρήσεων στην κοινή μας θάλασσα για λόγους οικονομικής απόδοσης, αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας. Τέλος, με πρότασή μας διασφαλίζεται η δημόσια χρήση παράκτιων ε, και θαλάσσιων περιοχών, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, για το κοινό, για ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Δανέλη. Απλώς να ειδοποιήσω τους ομιλητές μας ότι έχουμε ξεπεράσει το του χρόνου. Εάν δεν σεβαστείτε εσείς τα όρια, δεν θα μπορέσω και εγώ να σας δώσω τον λόγο. Κύριος Κύριε Πρόεδρε, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσουν εργαλεία για την ανάπτυξη τη δημιουργία θέσεων εργασία και την εκπλήρωση των στόχων τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Η Ένωση, ιδιαίτερα σε αυτέ τι δύσκολε εποχέ τη κρίση, χρειάζεται να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τη θάλασσα, που απασχολούν 5 εκατομμύρια άτομα και αποφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προστιθέμενη αξία τη τάξη των 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συντονισμό των διαφορετικών δράσεων τη θαλάσσια πολιτική σε πολιτικό επίπεδο, ώστε να βελτιστοποιήσουμε τα ωφέλη που απορρέουν για τα κράτη-μέλη και του Ευρωπαίου πολίτε. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζω την έκθεση τη συγγήτρια κυρία Μάισνερ για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη θεωρώ μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Για την ύπαρξη ενό ευρωπαϊκού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού είναι απαραίτητο η Ένωση να κινηθεί προ την κατεύθυνση του ελέγχου, τη σταθερότητα και τη ασφάλεια των παράκτιων και χωρικών υδάτων, των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τελειώνω κύριε Πρόεδρε, των υφαλοκρηπίδων, των αυτιλιακών υποδομών και των θαλάσσιων πόρων των κρατών μελών της Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα Σας ευχαριστούμε κύριε Σαλαβράκο, κύριε Κερμπάνκη. Για ένα λεπτάκι. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πρέπει να μεταρρυθμιστεί επιγόντως πολιτική αλίας. Ε, κατά σύστημα αλλιεύουμε περισσότερα από όσα αντέχει το οικοσύστημα. Υπάρχει λοιπόν υπεραλίευση. 80% των αποθεμάτων στη Μεσόγειο και 74% στον Ατλαντικό ε, υπεραλλιεύονται. Θα ήθελα λοιπόν να τα δω λίγο από τη σκοπιά της Ουγγαρίας. Κοιτάξτε, εμεί δεν έχουμε θάλασσα, οπότε δεν ξέρω γιατί μιλάω εγώ για την αλληλεία, αλλά πρέπει να γίνει η αλληλεία με τρόπο οικολογικό. Στόχοι τώρα τη μεταρρύθμιση. Στόχο είναι να έρθουν σε ένα βιώσιμο επίπεδο ξανά τα ήχθη αποθέματα και να μπορεί να τρώει και κανένα ψαράκι ο Ευρωπαίος πολίτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Mr. especially for speaking κύριε Μπάνκε, κυρίως που σεβαστήκατε τα όρια του χρόνου. Ο κύριος Καρόνα τώρα. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, και εγώ θα διαβάσω αυτά που προτιμάσα. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν ήθελα το Ευρωκοινοβούλιο να προδώσει τα όσα είπε μισή ώρα πριν στη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση τη πολιτική αλεία. Είπαμε ότι χρειαζόμαστε μια βιώσιμη πολιτική και να βοηθήσουμε τη θάλασσα για να παράγει περισσότερα. Μην προδώσουμε λοιπόν αυτήν την δέσμευση ε, εδώ. Θέλουμε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων αλλά και μια συνεπή θέση από το Κοινοβούλιο. Κανείς δεν ανησυχήσε όταν στη Μεσόγειο υπήρχε ε, η δυνατότητα για παρασυρώμενα δίχτυα σε χίλια μέτρα ε, βάθος. Εδώ πρέπει να δείξουμε την ίδια συνέπεια και προσοχή. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε κάτι για ένα μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτι άλλο για άλλε θέλωσε. Τρει προεδρίε, η Ιρλανδική, η Κυπριακή και η Λιθουανική, δεν προέλεψαν στι προτεραιότητέ του αυτό το θέμα. Και αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικά σοβαρό. Δεν θέλουμε να πούμε ότι υπήρξε μοναδράνη από αυτέ τι προεδρίε, αλλά υπήρχε και πρόθεση από τι ομάδε λόμπι για να προωθήσουν τα δικά του συμφέροντα στο Βόρειο Ατλαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καρόνα. Κλείνουμε τον κατάλογο των αγορητών και τώρα περνάμε στη διαδικασία κατευθείαν. Έχω πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά τίματα για αγόρευση. Δεν μπορώ να, δεχτώ, να τα δεχτώ όλα. Θα δεχτώ μόνο τρία. Πολλοί είναι που ήθελαν τον λόγο, δεν μπορώ να το δώσω δυστυχώ. Η κυρία είναι ο κύριο Μπορονίνη, η κυρία Φασίκοβα. Η κυρία Κάινεν Έχετε ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, υπάρχει υπεραλία, κάποιοι γόνοι ψαριών οριμάζουν πάρα πολύ αργά και δεν αυξάνονται ειδικά ε, δε τα μικρότερα είδη καρχαριών κινδυνεύουν από αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό πέρα από τις ε, τράτες ε, έγινε άλλη μια προσθήκη όσον αφορά τα είδη τα οποία κινδυνεύουν. Τα επιστημονικά στοιχεία επίσης ε, είναι σαφή. Όμως πάρα πολλοί στο Κοινοβούλιο θεωρούν πως έτσι θα επηρεαστεί ε, το βιός των ψαράδων και δεν θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. έπρεπε να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών ε, στόχων. Δηλαδή, εάν θα επηρεαστούν αρνητικά οι ψαράδες, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. Πρέπει όμως να δούμε ποιες είναι και οι εναλλακτικές. Παραδείγματο χάρη η Νορβηγία χρησιμοποιεί μια άλλη μέθοδο πολύ πιο φιλική προς τα ψαρία. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Μπονανίνη. Ένα λεπτό έχετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι αρνητικέ συνέπειε. Με συγχωρείτε. συγχωρείτε. Θα ήθελα να παρακαλέσω του ομιλητέ μα, αν μπορείτε να σηκώνεστε. Ξαναρχίζω. Οι αρνητικέ συνέπειε τη αλεία με παρασυρωμένα δίχτυα σε βαθαία ύδατα είναι ανυπολόγιστε καταστρέφονται αναπανόρθωτα οικοσυστήματα που είναι καθοριστικά για την παραγωγή ε, των ε, αληφτικών αποθεμάτων. Στατηγικές συνιστώσεις της συντήρησης των οικοσυστημάτων. Χάνουμε όλο και περισσότερο τον πληθυσμό των οικοσυστημάτων στη θάλασσα και την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα που προσφέρει θα πρέπει να προσέξουμε να μην υπερεκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα με τις ελληνικές μας δραστηριότητε, διότι οι αρνητικές συνέπειες που πλήττουν ένα οικοσυστήμα ε, στη συνέχεια περνάνε και στα γειτονικά. Η αλία με τα παρασυρώμενα δίχτυα έχει σοβαρές συνέπειες για τις ε, περιοχές όπου μπορεί να υπάρχει τέτοια δραστηριότητα. Θα πρέπει εδώ να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε μια αλληλευτική πολιτική που να είναι βιώσιμη, ώστε οι παράκτιες κοινότητες να στηριχθούν. Με συγχωρείτε που ξεπέρασα το χρόνο μου. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Δέχομαι τη συγγνώμη σας.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 κάποιων ε, ψαριών. Έχουμε κάποια είδη τα οποία χαρακτηρίζονται από πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το άλλο ζήτημα είναι πως η μέθοδος ε, αυτή με τις στράτες ε, εισήχθη πριν μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την επίπτωση στο οικοσύστημα μέχρι το 2003 δεν υπήρχε καμία ρύθμιση της μεθόδου αυτής ε, στα περισσότερα κράτη-μέλη. Οπότε πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση για να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε με τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Ε, η ψηφοφορία θα γίνει αμέσως μετά το επόμενο θέμα, το οποίο είναι... Η έκθεση Γκάρτια Θάμπαλ για τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προπολογισμό 2015. Δίνω τον λόγο αμέσως στην κυρία Γκάρτια Θάμπαλ. Για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι